σε μια σύντομη παρουσίαση της ακόλουθης έκθεσης των κυρίων, της κυρίας Ντανόκα και Μπλίνκεβιτσιούτε για τι συνθήκε ε, στην εργοεργασία που ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή και θα δώσω το λόγο στι συνεισηγήτριε για τέσσερα λεπτά η καθεμία. Ξεκινούμε με την κυρία Colleagues, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Η έκθεση την οποία έχετε μπροστά σας προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα στην κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη το ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τις ίδιες αμοιβέ και πρέπει να έχουν τις ίδιες αμοιβέ και τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες ευθύνες. Ο συνδυασμός νομοθετικών και μη μέτρων πρέπει να επιτρέψει τους άνδρες και τις γυναίκες να συνδυάσουν καλύτερα την φροντίδα των συγγενών τους, την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο τους και την προσωπική τους ανάπτυξη η αγορά της εργασίας δεν είναι σε θέση να παρέχει σε κατάλληλο επίπεδο ευκολίες σε σχέση με την εκμετάλλευση του χρόνου και αυτό έχει υψηλό κόστος για τους εργαζομένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές εξισορρόπησης της πραγματικότητας στον τομέα της εργασίας και της οικογενειακής ζωής σε μια κοινωνία η οποία αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ορισμένες νομοθετικές προτάσεις ε, για τις γονικές άδειες, να αναθεωρηθεί η οδηγία για τη γονική άδεια, όπως επίσης και να υπάρξει και μια οδηγία ειδική για αυτούς οι οποίοι φροντίζουν μέλη της οικογένειας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους αναπήρους, μέλη της οικογένειας και τους ασθενείς. Ένα ειδικό τμήμα της έκθεσης αφιερώνεται στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης. Σημειώνουμε επίσης και την αύξηση των εργαζομένων πτωχών όμως, που πρέπει να συνδυάζουν πολλές μορφές ενασχόλησης, απασχόλησης μάλλον, για να τα βγάλουν πέρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ικανοποιητική αμοιβή για όλους τους οργαζομένους και να υπάρχουν, όπως είπα, διευκολύνσεις στο ωράριο εργασίας που να μην δημιουργούν επιπλέον προβλήματα ε, και στους άνδρες και τις γυναίκες. Θα πρέπει επίσης ε, να εξισορροπηθεί όπως είπαμε η εργασία και η οικογενειακή προσωπική ζωή λαμβάνοντας υπόψη την διασφάλιση ε, των εργαζομένων έτσι ώστε να έχουν αρκετό χρόνο και για ξεκούραση και για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Οι συνεισηγητές λοιπόν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τις προτάσεις της ε, τελικής μας πρότασης. Είμαστε όμως ε, ε, ανήσυχες διότι έχουν ζητηθεί πάρα πολλές και χωρισμένες ψηφοφορίες, κατά διέρεση ψήφι δηλαδή. Και ιδιαίτερα σε σχέση με τα 11 δίκτυα των ΜΚΟ που συνεργάζονται από το 2012 έτσι ώστε να βοηθήσουν στην συνειδητοποίηση ε, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες στα πλαίσια της προσπάθειας να εξισορροπήσουν με σωστό τρόπο την εργασία και την οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να ψηφιστεί πλήρως η πρότασή μας έτσι ώστε να μην υπονομευθεί ε, το νόημά του. Παρακαλώ μην αγνοήσετε το συγκεκριμένο αίτημα. Η Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την συνεισηγήτρια διότι είναι σημαντικό. Ευχαριστώ την κυρία Σντανόκα και όλους και όλες που συνεργάστηκαν για αυτή την έκθεση. Είναι αυτή η έκθεση η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποφάσεις και συστάσεις που θα βοηθήσουν να συνδυαστεί η επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή, ιδιαίτερα για οικογένειες με παιδιά και σε σχέση και με τη δημόσια διαβούλευση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα θέματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και προσδοκούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πληρέστερες ε, προτάσεις ε, ε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Τον Ιούνιο εφέτος υιοθέτησε τις συστάσεις του το Συμβούλιο για την ισότητα των φύλων συνιστώντας την ενίσχυση, την ενδυνάμωση νομικών μέτρων ώστε να μπορέσει να συνδυαστεί καλύτερα για τις γυναίκες και τους άνδρες η επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή. Είμαστε όλοι αυτούς τους στόχους. Γι' αυτό ζητούμε να υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γονεϊκή άδεια. Επίσης, σε σχέση με την δημιουργία όρων και προϋποθέσεων, ώστε να μπορούν να διασφαλίζονται τα άτομα που χρειάζονται, που χρήζουν φροντίδας και μέρημνας στις οικογένειες και ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία πρόταση για την πατρική άδεια σε σχέση με επαρκή χρονικό διάστημα για τους ε, πατέρες και επίσης να υπάρξει μια σύσταση που θα επεκτείνει από τέσσερις σε τουλάχιστον έξι μήνες αυτή τη διάρκεια αυτής της άδεια. Οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Είναι θεμελιώδες ε, ζήτημα για τις γυναίκες. Ένα θέμα είναι να μπορούν οι, εργα... οι γυναίκες να εργάζονται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυτό απαιτεί να προσαρμοστούν εφαρμόσουμε τις δυνατότητες ε, της επαγγελματικής ζωής των γυναικών ώστε να μπορούν να συνδυάζονται και να ταιριάζουν με τις οικογενειακές ανάγκες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη γερνά, ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά ταχύτατα. Γι' αυτό οι οικογένειες θα πρέπει να έχουν περισσότερο χρόνο να μπορούν ε, να περάσουν με τα μέλη, με τους οικείους τους, με τους συγγενείς τους ε, στο σπίτι τους, στον οικογενειό τους ε, δεν είναι το θέμα του αν θα μπορεί κανείς να έχει περισσότερα ή όχι παιδιά όταν δεν υπάρχουν οι πιο θετικοί όροι και προϋποθέσεις για να φέρει κανείς παιδιά στον κόσμο και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φθήνουσας δημογραφικής εξέλιξης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την απασχόληση των γυναικών ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα οικογενειών με παιδιά. Ευχαριστώ. Επίση, θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη την, τον συνδυασμό και την ε, δυνατότητα να μπορούν να ταιριάζουν την επαγγελματική με την οικογενειακή του ζωή γυναίκες και την ε, δυνατότητα να επικεντρωνόμαστε στις ε, αναγκαίες συνθήκες για την φροντίδα των παιδιών και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους στόχους που πρέπει να επιτευθούν για να μπορέσει η οικογενειακή ζωή να ταιριάξει καλύτερα στις ανάγκες των οικογενειών. Δεν υπάρχει μία λύση για όλους ισοπεδωτικά. Πρέπει να δούμε τις ειδικέ ανάγκες των οικογενειών. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι από τις διαφορετικές πολιτικές ομάδες κατανοούν την σπουδαιότητα αυτού του ζητήματος και πρέπει να αποστείλουμε και ένα σαφές μήνυμα ότι έχουμε κατανοήσει τα προβλήματα που υφίστανται και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε και με τις προτάσεις αυτές θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Φτάνουμε τώρα στη δικασία του Catch Κύριε Σόιντοβα πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της δύο συναδέλφους. Έχει σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει το θέμα αυτό λόγω των αρνητικών δημογραφικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, γιατί υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στις προσπάθειες μιας πολιτικής για την οικογένεια που να επιτρέπει την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των πολιτών. Επίσης θα πρέπει να διευκολύνεται έτσι ώστε να υπάρχουν υπηρεσίες που θα φροντίζουν τα μέλη της οικογένειας που έχουν ανάγκη εφόσον οι υπεύθυνοι της οικογένειας οφείλουν να εργάζονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει και κάποιες δομές οι οποίες έχουν ε, σαν στόχο να αντικαταστήσουν τις οικογενειακές δομές και αυτό δεν είναι καλό βέβαια. Um, I'd like to thank my... Θέλω να ευχαριστήσω τις ε, δύο συναδέλφους για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν είναι πολύ σημαντικό η έκθεση να λάβει σαφή θέση κατά της λιτότητας και υπέρ της ισότητας. Υπογραμμίζει την θλιβερή πραγματικότητα ότι οι γυναίκες είναι αυτές που πλήττονται από τις περικοπές κατά βάση. Η Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση βάσει αυτών που αναφέρεται εδώ η έκθεση. Η προώθηση των ισοτήτων ε, της ισότητας μεταξύ φίλων είναι πολύ σημαντικό και αυτό, πάνω σε αυτό στηρίζονται οι βασικές αξίες της Ένωσης. Εμείς ε, έχουμε ευθύνη να υπογραμμίσουμε τη σημαντική δουλειά που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, εξασφαλίζοντας ότι οι ψηφοφόροι μας στη Βρετανία θα συνεχίζουν να προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προστασία των Παιδιών σε κάθε περίπτωση. Ο κ. Μαριάς. που έχουν αναλυφθεί μέχρι στιγμή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την εξισορρόπηση τη επαγγελματική και προσωπική ζωή, δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα, οι διακρίσει που παρατηρούνται στου εργασιακού χώρου ανάμεσα στα δύο φύλλα καθιστούν για τι γυναίκε ακόμη πιο δύσκολη την εναρμόνιση αυτή οι τύποι αδεία που συνδέονται με οικογένειακού λόγου, εξακολουθούν να επιφέρουν δυσμενείς διακρίσεις παρά την υφιστάμενη νομοθεσία ενώ σε χώρε όπω η ελλάδα οι έντονε μισθολογικέ διαφορέ και τα ποσοστά ανεργία που φτάνουν στο 28,7 στι γυναίκε, τι καθιστούν οικονομικά ευάλωτε. Επομένω, είναι αναγκαίο η ένωση να αναλάβει πολιτικέ δράσει προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικο οικονομικέ προκλήσει που δημιουργούνται στα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο όσο εξακολουθούν να επιβάλλονται πολιτικές λιτότητας στι ευρωπαϊκές χώρες του νότου η εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματική ζωής καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη θα γίνονται ακόμη πιο δύσκολες. ευχαριστώ. Κύριος Γιάκοψιτς. Ευχαριστώ Πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασε η Εκπληξίζω όταν είδε ότι ζήτησα το λόγο. Ξέρετε, συχνά έρχομαι στη διαδικασία του Κατζηράη. Αυτή τη φορά όμως θέλω να σας πω την εμπειρία μου. Έχω 25 χρόνια στην πολιτική σε μια συντηρητική χώρα όπως είναι η Κροατία. Προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ισότητα των φύλων και κατά της ε, των διακρίσεων και στην αγορά εργασία και στην πολιτική. Όταν κατα... έκανα λοιπόν τον, το, το, τους εκλογικούς καταλόγους ε, των υποψηφίων του κόμματος μου, προσπαθούσα πάντα να υπάρχει μια ισορροπία για να έχουμε... και πάντα έβαζα μια γυναίκα περισσότερο στο συνδυασμό. Αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ένα θετικό μήνυμα. Θα ευχόμουν κι εγώ πολλοί άνδρες να λάβουν το λόγο ε, για το θέμα αυτό. Ο κύριος Λόπες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την επιβολή πολιτικών λιτότητας ε, και η εκμετάλλευση που ακολουθούν οι κυβερνήσεις ε, δημιουργούν οπισθοδρομήσεις ε, κοινωνικές που πλήττουν ιδιαίτερα τους στοχούς. Έχουμε 30 εκατομμύρια άνεργους και όλο και μεγαλύτερη αδικία στην κατανομή του πλούτου. Βλέπουμε εδώ και ε, την επίθεση κατά των κοινωνικών πολιτικών. Βλέπουμε την υποβάθμιση των μισθών, τον επισφαλή χαρακτήρα της εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα και για την οδηγία για την γονεϊκή άδεια δεν ε, ανταποκρίνονται τα πράγματα στις ανάγκες. Πολιτικές ε, που τώρα προσπαθούν κάποιοι να συγκαλύψουν ε, με την επίκληση των κοινωνικών θεμάτων και βλέπουμε εδώ ότι αυτά θα γίνουν μόνο εφικτά όταν θα υπάρξουν οι σωστές πολιτικές για την υποστήριξη των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Ούρτασουν. Ο κύριο Σεμπαστιαν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Είναι σαφή η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη να συνδυαστεί καλύτερα η οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Χρειάζονται αποφασιστικά και σωστά μέτρα. Τα είπε ο Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα ε, δεν ε, επιτυχάνει και τέτοιο. Κρύβει αυτά που έχουν συμφωνηθεί, όπως ε, το αίτημα για ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο για την γονική άδεια. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση αυτή, στην διαδικασία της Επιτροπής δεν θα υπάρξει ποτέ μια πραγματική εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κάτι που είναι θεμελιώδες επαναλαμβάνω για τις στρατηγικές της ισότητας και που περιλαμβάνονται σε όλες τις συνθήκες της Ένωσης. Δεν θα είναι δυνατόν αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, αυτός ο πολιτικός προσανατολισμός. Ευχαριστώ. Κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο Πρόεδρε. Και εγώ βλέπω ορισμένες θετικές πλευρές στην έκθεση. έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και κάποια αρνητικά σημεία. Οι εργασιακές διατάξεις περιλαμβάνουν ε, ορισμένα στοιχεία τα οποία καθιστούν την ομοθοσία δίσκαμπτη και πατερναλιστική. Εδώ είναι θέμα θα έλεγα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων ή ίσως και συλλογικών διαπραγματεύσεων και όσοι ε, εργάζονται στην αγορά θα πρέπει να εργάζονται σύμφωνα με τους κανόνες ε, της επικουρικότητας και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι κυρίαρχα στον συγκεκριμένο τομέα. Η κυρία Αρενά. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στα συνδικάτα. Θα ήθελα να πω ότι παρά τα αιτήματα των συνδικάτων και των εθνικών συνδικάτων και του Ευρωπαϊκού Συνδικάτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 αποφάσισε να εγκαταλείψει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γονική άδεια λέγοντας ότι η οδηγία αυτή δεν ήταν σύγχρονη και δεν άνοιξε τις ε, δυνατότητες συνδυασμού ε, της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή. Ευχαριστώ τις δύο συνεισηγήτριες. Είναι μια σύγχρονη και πλήρης έκθεση. Ε, Προτείνουν μια νομοθετική αντιμετώπιση των γονεϊκών αδειών και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Αυτό είναι σύγχρονο Προτείνει επίσης μία εγγύηση για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να γίνουν δεκτά σε δομές υποδοχής έτσι ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της φτώχειας και προτείνει η έκθεση αυτή ότι όλα αυτά θα πρέπει να εγγραφούν στα θεμελιώδη δικαιώματα, στα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι μια σύγχρονη έκθεση και ευχαριστώ τις συνεισηγήτριες. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις δημογραφικές αυτές αλλαγές. Το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής οδηγεί σε χαμηλότερη γεννητικότητα. Υπάρχουν αυτές οι μεταβολές, υπάρχουν νέοι συσχετισμοί όσον αφορά την κοινωνία και υπάρχουν και τα μεταναστευτικά ρεύματα και πρέπει να δούμε πώς θα ακολουθηθούν πολιτικές που θα μπορέσουν να συμφιλιώσουν την εργασιακή ζωή με την οικογενειακή ζωή. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών ώστε να εκπονηθούν οι σωστές πολιτικές για την υποστήριξη πολιτικών κατά της δημογραφικής φθήνουσας πορείας και για την υποστήριξη μεγαλύτερης συνοχής στις οικογένειες. Ευχαριστώ τις εισηγήτριες για αυτήν την έκθεση που αναφέρει σημαντικά στοιχεία για την συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η προσπάθεια εξισορρόπησης της προσωπικής ζωής με την επαγγελματική ζωή είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Οι νέοι αναγκάζονται να κάνουν πολλές δουλειές για να ισορροπούν τα οικονομικά τους και τα οικονομικά των οικογενειών τους. Οι συνθήκες απασχόλησης είναι όλο και πιο δύσκολες. Εγώ έχω εργαστεί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ο κόσμος ε, χρειάζεται περισσότερη δουλειά αλλά κυρίως χρειάζεται περισσότερο χρόνο οι εργοδότες πιέζουν θα έλεγα τους εργαζομένους οι οποίοι με τη σειρά τους πιέζουν την προσωπική τους ζωή και δεν έχουν μια εξισορροπημένη προσωπική δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν μονομερώς οι εργοδότες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι φιλόδοξη, και να ισορροπεί την προσωπική ζωή και την επαγγελματική ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με το Catch the Δίνω το λόγο στον κύριο Επίτροπο. Ο κύριος Τσίλιανιδης, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος των αγαπητών συναδέλφων μου επιτρόπων Μάριαν Τάισεν και ε, κυρία Γιούροβα τις δύο συνεισηγήτριες την κυρία Σντάνουκα και την κυρία Μπλίνκεβιτσούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται πολλά από τα στοιχεία των αναλύσεων που παρουσιάσατε και των συμπερασμάτων σας θα πρέπει γενικότερα η φροντίδα και η μέρημνα να μην θεωρείται μόνο αποκλειστική υπόθεση των γυναικών εφεξής, Το να προσέχει κανείς και να φροντίζει είναι δουλειά οποιοδήποτε σήμερα. Πολλοί θα ήθελαν να έχουν περισσότερο χρόνο για να περάσουν με την οικογένειά τους και να μην υπάρχουν προσκόμματα και εμπόδια που θα τους αποθαρρύνουν να το πράξουν. Θεωρεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν στοχεύουμε στο να ε, υπάρχει μεγαλύτερη ενεργητικότητα και δράση στην αγορά εργασίας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τις γυναίκες να απασχοληθούν και να δράσουν στην εργασιακή ζωή και το αποφασίσουν αν θα έχουν παιδιά ή όχι ή αν θα ε, δράσουν με τον ένα ή άλλο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για έναν εργαζόμενο άνδρα ο οποίος θα επιθυμούσε να είναι περισσότερο χρόνο στο σπίτι του ώστε να ασχοληθεί περισσότερο με τα παιδιά του όσο είναι μικρά ή και με τους συγγενείς τους που χρήζουν υποστήριξης και βοήθειας. Είναι λοιπόν ε, εύκαιρη αυτή η έκθεση για την, ε, στο συγκερασμό και τη συμφιλίωση εργασιακής ζωής με την, με την οικογενειακή ζωή ώστε να μπορέσει να, να τύχει προσοχής το θέμα των σημαντικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να προταθούν συγκεκριμένες δράσεις. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να παρουσιάσει τώρα μια πιο σφαιρική, ολιστικού χαρακτήρα δράση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Έχουμε ήδη έργο στον τομέα αυτό όπως τις κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, benchmarks, βέλτιστες προδιαγραφές αλλά όλα αυτά δεν επαρκούν. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και τα νομικά μέσα και τα μέσα πολιτικής πρέπει να εξυγχρονιστούν, να επικαιροποιηθούν και να είναι πιο αποτελεσματικά. Πρώτον, για να δίνεται η δυνατότητα και σε άνδρες και σε γυναίκες να δραχθούν της ευκαιρίας να ενδυναμώσουν το δυναμικό τους στην αγορά εργασίας και να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι στο να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και τέταρτον να μειωθεί η έκθεση με βάση το στην φτώχεια και να επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ των φύλων. Μέσα σε ένα σφαιρικό ευρύτερου χαρακτήρα πακέτο μέτρων που θα υποστηρίζει τους στόχους αυτούς για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους γονείς ξεκινούν όταν ε, αποκτούν ένα παιδί ε, στην οικογένειά τους και πρέπει να υπάρχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο φροντίδας παιδιών από πλευράς υποδομών που θα διασφαλίζονται ώστε να έχουν τη σωστή επιλογή οι ε, πολίτες και να μην ξεχνάμε και την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την φροντίδα που πρέπει να την χάνουν ηλικιωμένοι ή εκείνοι που, πρέπει, που χρήζουν βοήθειας στις οικογένειες. Προτείνουμε λοιπόν, θα προτείνουμε επικαιροποιημένες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπιστούν οι ε, ε, ανάγκες όπως υφίστανται. Περνάμε τώρα στη δεύτερη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Αναζητούμε τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για το νομοθετικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια ευρύτερη διαβούλευση που διεξήχθηκε που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος είναι ένα άλλο στοιχείο. Επίσης οι απόψεις που εκφράστηκαν όσον αφορά από τους κυριότερους εμπλεκόμενους για την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολόκληρου ε, εύρους μέτρων μη νομοθετικού χαρακτήρα για παράδειγμα όπως συστάσεων βελτιωμένης εποπτείας καλύτερης χρήσης κονδυλίων και κοινών δράσεων υπό τις, ε, τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων μέσα στο πλαίσιο αυτό πρόθεση της Επιτροπής είναι να συνοδεύσει όλες αυτές τις δράσεις δραστήρια. Σε περίπτωση που κοινωνικοί εταίροι αποφασίσουν να μην προβούν σε διαβουλεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στο να εξετάσει όλες τις δυνατότητες για την ε, κατάληξη σε μια αποτελεσματική πολιτική. Είδατε αυτή τη δέσμευση στο πρόγραμμα εργασίας μας και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα βιώσουμε, θα ζήσουμε την υποστήριξη από πλευρά σας ε, προς αυτή τη φιλοδοξία ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις από κοινού προς όφελος των γυναικών και ανδρών που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Προχωρούμε τώρα τις ε, παρεμβάσεις ε, του ενός λεπτού βάσει του άρθρου 163 του κανονισμού. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο